δεν είχαν καθόλου χρόνο αγόρευσης και δόξατε ε, catch the eye, δώσατε χρόνο αγόρευση σε άλλες ομάδες πολιτικές που είχαν πάρει επανειλημμένα το λόγο πριν ενώ στους μία δεν δώσατε το λόγο.